αξιότιμη ε, πρόεδρε των πολιτικών ομάδων, κύριοι Ευρωβουλευτές, ε, κυρίες μου. Είναι μεγάλη τιμή μου να απευθύνομαι στο κοινοβούλιο αυτό, διότι όταν είχα έρθει τον Ιανουάριο τέλωσα την ομιλία μου λέγοντας ότι η οικονομική κρίση έθεσε σε μεγάλη δοκιμασία την Ευρωπαϊκή Ένωση και τώρα πρέπει να κάνω τον απολογισμό της Δανικής Προεδρίας σε μια μεγάλη περίοδο κρίσεως της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και υπάρχει μία πρόκληση την οποία αντιμετωπίζει η Ένωσή μας και δεν πρέπει να την υποτιμήσουμε. Το είπα ήδη στην αρχή της Προεδρίας μας. Όχι ε, χωρίς να γνωρίζω τι ε, θέλατε από την Δανική Προεδρία αλλά για να προσδιορίσω τι διακυδεύεται εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να επιλύσει αυτή την κρίση. Τους τελευταίους μήνες χρειάστηκε να λάβουμε σημαντικές αποφάσεις ε, για να τοποθετήσουμε τις βάσεις του ευρώ για το μέλλον και αυτό δεν είναι κάτι το εύκολο σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση πολλών διαφορετικών και ποικίλων πτυχών όπως η δικιά μας. Ποτέ όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση σήματα, την οικονομική βάση, το, τη μελλοντική ευημερία, τα όνειρα και τις προσδοκίες των παιδιών μας δεν έχει περάσει ακόμη η μπόρα και ακόμη αντιμετωπίζουμε πολλά δύσκολα ε, προβλήματα και πολλές ε, ε, προκλήσεις. Ελπίζω λοιπόν ότι μπορώ να εμπνευστώ από τα λόγια του Κόντρα Τάντενάουερ του πρώτου καγκελαρίου της, της Γερμανίας που είπε ότι το όνειρο λίγων η Ευρώπη έγινε η προσδοκία πολλών και τώρα έγινε η πραγματικότητα για όλους Ποτέ αυτά δεν ήταν τόσο σωστά όσο σήμερα. Η Ευρώπη είναι ανάγκη για όλους μας. Και ε, σαν εκπρόσωπος των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων έχουμε και αισθανόμαστε μία υποχρέωση να βρούμε μία λύση η οποία θα προχωρήσει την Ευρωπαϊκή μας Ένωση και το οφείλουμε στους πολίτες μας. Όταν στεκόμουν μπροστά σας τον ε, Ιανουάριο είπα ότι κατά βάση ε, και στην καρδιά μου είμαι Ευρωπαία και στους τελευταίους έξι μήνες επιβεβαιώθηκε η πίστη μου στο ευρωπαϊκό εγχείρημα. Πιστεύω ότι έχουμε κοινέ ευθύνε και κοινού στόχους. Εάν προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε την αλληλεγγύη, την ανάπτυξη και την ευημερία θα πρέπει από κοινού να επιζητήσουμε ε, να βρεθούν λύσεις και αυτή, αυτός θα είναι και ο στόχος της ε, Προεδρίας μας να, να εξασφαλίσουμε από κοινού αλληλεγγύη, ανάπτυξη και ε, πρόοδο. Ελπίζουμε ότι μπορούμε να ε, δώσουμε τους αναγκαίους πόρους εις τους πολίτες και αυτό βασίζεται σε έμπνευση κάποιο το οποίο τιμούμε, ο οποίος είχε πει το 1950 ότι η Ευρώπη δεν θα γίνει με τις μιας ή μόνο με ένα πρόγραμμα θα γίνει ε, βάση απτών επιτευμάτων που θα βασίζονται καταρχήν στην ελληνική. Ο Ρομπέρ Σουμάν το είχε πει αυτό και η ιστορία μετέπειτα της Ευρώπης απέδειξε ότι είχε απόλυτο δίκιο. Πιστεύω ότι υπάρχει αδιαφυσβήτητη αλήθεια στο θέμα αυτό. Η Ευρώπη βασίζεται ε, από ε, τα θεμέλια της ε, σε τουβλάκια αλληλεγγύης. Ορισμένα ήταν μικρά, άλλα μεγαλύτερα και βάσει αυτών των τουβλών οικοδομήθηκε η ανάπτυξη και η πρόοδος και αυτή είναι η ουσία της ε, Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αυτό προσπαθούμε να εργαστούμε βήμα προς βήμα και να επιτύχουμε αποτελέσματα. Να αναλάβουμε τις οικονομικές μας ευθύνες, ε, να έχουμε μία πιο πράσινη Ευρώπη. Ε, αυτή είναι μερική από τους στόχους της, Ευρωπαϊ... της Δανικής Προεδρίας. Αλλά δεν πρέπει να μείνουν τα λόγια χωρίς ουσία και ελπίζω ότι τον τελευταίο μήνα κάτι πετύχαμε το σύμφωνο για την ανάπτυξη και την απασχόληση είναι ένα επίτευγμα της Προεδρίας. Δεν θα λύσει όλα τα προβλήματα της Ευρώπης, αλλά είναι ήδη ένα φως στο σκοτάδι για πολλούς Ευρωπαίους πολίτες οι οποίοι αισθάνονται τις δυσχέρειες της ευρωπαϊκής κρίσεως. Για αυτούς που είναι εκτός της ε, αγοράς εργασίας, που δεν έχουν ευκαιρίες, που δεν έχουν καλές και ιδίω οι νέοι πρέπει να προσφέρουμε ένα βήμα προς τα εμπρός και ε, να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη. Βεβαίως η εργασία μας δεν τελειώνει εδώ, θα πρέπει να επαγρυπνούμε και να υλοποιήσουμε αυτό το σύμφωνο για να μπορέσει να αποτελέσει πρακτική πραγματικότητα, να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε και να πείσουμε τους λαούς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι μπορούμε να προχωρήσουμε βάσει αυτού του συμφώνου. Υπάρχει μια κατάσταση όπου για πρώτη φορά στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως δεν μπορούμε να προϋποθέσουμε ότι οι επόμενες γενιές θα έχουν περισσότερη ευημερία από ό,τι εμείς είχαμε στο παρελθόν και αυτό μας δίδει μεγάλη ευθύνη για τις συνθήκες των επιχειρήσεών μας και αυτή ήταν η προτεραιότητα της Προεδρίας μας. Θα ήθελα να αναφερθώ σε μερικούς από τους στόχους της Δανικής Προεδρίας. Με ζητήσαμε να υπάρξουν πιο ισχυρά μέτρα στο θέμα της έρευνας, της παιδείας, στην ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς για να υπάρξει ένα νέο λάκτισμα για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Χαίρομαι διότι επιτύχαμε να έχουμε έναν ιστορικό συμβιβασμό στο Συμβούλιο για την αναθεώρηση των διπλωμάτων ευρασιτεχνίας πράγμα το οποίο θα μειώσει το κόστος για όλες τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη ε, εξοικονόμηση η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Δεν έχουμε ίσως ακόμη όλα τα στοιχεία αυτού του συμβιβασμού αλλά ελπίζουμε ότι σαν ε, συν ε, νομοθέτες θα μπορέσουμε να εργαστούμε προς όφελος των εθνών μας. Επίσης ε, υπάρχει ένας νέος κανονισμός που θα μειώσει το κόστος της χρήσεως κινητής τηλεφωνίας και ε, το βάρος στις επιχειρήσεις και ελπίζουμε ότι και αυτό θα συμβάλλει στην ανάπτυξη. Επίσης υπάρχει ε, η ρύθμιση του θέματος τυποποίησεως για πρόθεση της ενιαίας αγοράς και ε, όσον αφορά τα κεφάλαια κινδύνου ελπίζουμε ότι θα υπάρξει πρόσβαση ε, για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες ε, στον κοινωνικό τομέα και θα προωθηθεί και εκεί η ανάπτυξη. Η ενιαία αγορά ήταν το μεγαλύτερο επίτευγμα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και θα πρέπει για να το προωθήσουμε να μεταρρυθμιστούμε και να εξυγχρονιστούμε. Ο δεύτερος δεύτερος βασικός στόχος της Προεδρίας μας ήταν να εξασφαλίσουμε μία πιο υπεύθυνη αγορά και ε, να την θωρακίσουμε εναντίον της οικονομικής κρίσεως του αύριο. Έχουμε λάβει σημαντικά μέτρα κατά την Προεδρία με τη συμφωνία για το 2 για τα δημοσιονομικά προγράμματα που εκπώνησε η Ευρωζώνη ζώνη για κοινού κανόνες που θα ενισχύσουν την εποπτεία και θα μπορέσουν να ε, εξισορροπήσουν τα μεγάλα πλεονάσματα και τα τεράστια χρέη. Είναι μερικούς από τους στόχους που είχαμε θέσει για την Προεδρία μας. Επίσης όσον αφορά τις κεφαλαιοχικές απαιτήσει ε, είχαμε προωθήσει τον κανονισ... την οδηγία η οποία θα εξασφαλίσει ότι δεν θα επαναληφθεί η κρίση που μας έπληξε το 2008. Τα κράτη-μέλη πρέπει επίσης να προωθήσουν διαρθρωτικές αλλαγές. Ολοκληρώσαμε το πρώτο εξάμεινο με ένα βασικό βήμα για μια πιο υπεύθυνη Ευρώπη. Όλα αυτά τα αποτελέσματα θα βοηθήσουν να αυξήσουμε την εμπιστοσύνη στο δημοσιονομικό πρόγραμμα της Ευρώπης και δεν αμφιβάλλω ότι το μήνυμα αυτό θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη υπευθυνότητα και μεγαλύτερη δημοσιονομική πειθαρχία Τέλος, έχουμε εργαστεί σκληρά για να δρομολογήσουμε τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό για να δημιουργηθεί ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό επίσης σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και γι' αυτό ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την επικοδομητική συνεργασία τους καθ' όλη την περίοδο. Είμαστε πεπισμένοι <clears throat> ακράδαντα ότι χρειαζόμαστε περισσότερους πόρους για την έρευνα, την παιδεία και την πράσινη τεχνολογία για να μπορέσει να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα τα οποία μπορούν να εξασφαλίσουν δημιουργία θέσεων εργασίας ήταν στόχος της Δανικής Προεδρίας κατά το εξάμεινο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το τόνισε και την περασμένη εβδομάδα. Όπως όλοι γνωρίζετε, η μετάβαση προς μία πράσινη οικονομία ήταν επίσης ένας βασικός στόχος της Δανικής Προεδρίας και χαιρετίζω τη συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε για την οδηγία για την πράσινη ενέργεια διότι χρειάστηκε μεγάλη ευελιξία, πολλή υπομονή και σκληρή εργασία και από τις δύο πλευρές. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω όλους όσους παρίστανται εδώ που συνέβαλα στην επίταξη αυτού του στόχου. Χωρίς εσάς δεν θα τα είχαμε καταφέρει. Και αυτή η οδηγία είναι πολύ σημαντική στην προσπάθειά μας επιτεύξεως του στόχους να δημιουργηθεί στην Ευρώπη μία οικονομία με ε, χαμηλό διοξίδιο του άνθρακος και πράσινη ανάπτυξη και επιπλέον η οδηγία αυτή θα δημιουργήσει εκατοντάδες χιλιάδες νέων θέσεων εργασίας στην Ευρώπη και θα εξασφαλίσουμε ότι η, Δανική, Ευρωπαϊκή Ένωση θα πλησιάσει τους στόχους που έχει θέσει για το 2020 αξιολογώ σαν εξαιρετικό το αποτέλεσμα αυτό. Θέλω να τονίσω την εκτίμησή μας για την αφοσίεση, την φιλοδοξία και την ευελιξία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την επίτευξη στόχων σε αυτή την μεταβατική περίοδο προς μία πράσινη οικονομία. Ο στόχος αυτός θα πρέπει να επιζητηθεί επίσης και τα επόμενα χρόνια για να μπορέσει να υπάρχει υπάρχει μία πιο πράσινη Ευρώπη και να εξασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη θα είναι ασφαλής. Η Προεδρία της Δανίας επέτυχε πολλά, πολλούς στόχους σε αυτό το τομέα και ε, αναγνωρίσαμε τη Σερβία σαν υποψήφια χώρα και ε, θα μπορέσουμε κατά αυτόν τον τρόπο να σταθεροποιήσουμε τα Δυτικά Βαλκάνια. Επίσης συμφωνήσαμε ε, στα θέματα του πακέτου ασύλου για να υπάρχει αποτελεσματικότητα, εξασφάλιση νομίμων δικαιωμάτων και καλύτερη συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Κυρίες και κύριοι, μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταφέραμε να καταλήξουμε σε πολλούς βασικούς τομείς και μπορώ να πω σήμερα ότι έχουμε επιτύχει ε, σημαντική ε, συμφωνία μόνο χάρη στην επικοδομητική συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κρατών μελών και Συμβουλίου. Ε, θεωρώ ότι οι στόχοι και τα επιτεύγματα της Δανικής Προεδρίας είναι και επιτεύγματα του Ευρωπαϊκού Ευρωπαϊκού Μπορέσαμε να υλοποιήσουμε ε, την ε, μέθοδο της Ευρώπης, έπαιξε ο καθένας το ρόλο του και σε ορισμένες περιπτώσεις ε, υπερμαχόμαστε αντικρουόμενα συμφέροντα. Η Ευρώπη δεν καλύπτεται όλοι από τις ίδιες απόψεις πάντοτε. Μπορέσαμε να προωθήσουμε τον μηχανισμό αξιολογήσεως και αυτό χαρακτηρίζει τις προσπάθειές μας. Υπήρξε όμως ευελιξία κατά το εξάμεινο, θέληση να επιτύχουμε έναν κοινό στόχο και μία αφοσίωση εις ε, ε, ε, στις ανάγκες και τους στόχους των πολιτών οπότε ένα-ένα τουβλάκι μπορέσαμε να προωθήσουμε το οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως προσπαθώντας λοιπόν να οθήσουμε την Ευρώπη προς ένα μελλοντικό στόχο ανάπτυξης θέλουμε να δημιουργήσουμε με την Ευρώπη που εμείς ονειρευόμαστε, της οποίας όλοι είναι μέλη και ε, είναι ένα μοναδικό οικοδόμημα. Αυτό πιστεύω, αυτό είναι που βοήθησε τις οικονομίες μας να είναι τόσο επιτυχής κατά τα προηγούμενα χρόνια και θα βοηθήσει να τις αναπτύξουμε και στο μέλλον διότι ε, το, η Ευρώπη πρέπει να προωθηθεί πέραν της ε, κρίσεως και αυτό δεν είναι θέμα του κοινωνικού μας προτύπου πρέπει όμως να μπορέσει η ε, Ευρώπη το επιτύχει να επιτύχει την αλληλεγγύη ε, φτιάχνοντας ε, δίχτυα ασφαλείας και δημιουργώντας ίσες ευκαιρίες για όλους. Οι δύσκολες αποφάσεις που λαμβάνουμε σήμερα, αύριο, δεν θα πρέπει να αποτελέσουν, ε, να, να οδηγήσουν σε απομάκρυνση από την αλληλεγγύη. Αντιθέτω, αυτό το κάνουμε για να προστατεύσουμε τον τρόπο ζωή μα, το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο μας, ε, τις αξίες μα και θα συνεχίσουμε να κάνουμε το ίδιο. Μόνο τρόπος για να προχωρήσουμε είναι στενότερη συνεργασία και ισχυρότερη συνεργασία μεταξύ όλων μα. Απάντηση στι ε, προκλήσει που αντιμετωπίζει η Ευρώπη είναι περισσότερη η Ευρώπη και όχι λιγότερη και αυτή ήταν η κατευθυντήρια αρχή για τη Δανέζικη Προεδρία καθ' όλη τη διάρκεια της. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την κυρία Τόνι Σμιτ. Τώρα εν ονόματι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το λόγο έχει ο πρόεδρος κύριος Μπαρόζο. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Πρωθυπουργέ, Αξιότιμοι κύριε Ευρωβουλευτέ, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία την Πρωθυπουργό ε, Σμιτ και όλη το επιτελείο τη, ιδιαίτερα τον Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων κύριο Σβάμεν, για μια πολύ δυναμική Προεδρία. Το πρόγραμμα της Προεδρίας ε, είχε τον τίτλο «Η Ευρώπη στη δουλειά». Ε, είναι δίκαιο λοιπόν να πει κανείς ότι και εσείς ήταν μια Προεδρία που δούλεψε σκληρά και κατεβάλλατε κάθε προσπάθεια για να συμβάλλετε στην ε, ευρωπαϊκή ολοκλήρωση σε αυτές τις δύσκολες ε, φάσεις. Ε, ιδιαίτερα προσωπικά θα ήθελα να σας ευχαρώ για την ετοιμότητά σας και για την δέσμευσή σας στην πράσινη ατζέντα. Ε, τομέα στον οποίο η Δανία αποτελεί μεγάλη έμπνευση και υπόδειγμα, όχι μόνο για την Ευρώπη αλλά και για τον υπόλοιπο κόσμο. Όλα αυτά αντικατοπτρίζονται και στα πορίσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που καλύπτουν το, πλήρη, το πλήρες φάσμα των ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων. Εφώς, ε, από τότε που συζητήσαμε την τα πορίσματα αυτά αμέσω μετά από τη διάσκεψη κορυφή. Εδώ θα τονίσω μόνο συγκεκριμένα ζητήματα. Θα ξεκινήσω με την οικονομία. Σχεδόν ολοκληρώθηκε το δεύτερο ευρωπαϊκό εξάμεινο. Σοβαρή και ει βάθο εργασία έχει γίνει επί τη βάση των προτάσεων τη Κομισιόν για συγκεκριμένε συστάσει για κάθε χώρα. Εγώ είμαι ικανοποιημένο με τη συνένεση που προκύπτει γύρω από αυτέ τι συστάσει. Αυτή η εργασία φυσικά δεν μπορεί να διαχωριστεί από την ατζέντα μας για την οικονομική ανάπτυξη. Όπως κατέστησε σαφές η Κομισιόν, η ανάπτυξη μπορεί μόνο να επιτευχθεί μέσω του συνδυασμού διαρθωτικών αλλαγών και στοχευμένων επενδύσεων και τώρα γνωρίζετε αυτό μέσω της Δανέζικης Προεδρίας και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για αποφασιστική δράση υπέρ της ανάπτυξης. Επίσης είμαι ικανοποιημένο με τον τρόπο με τον οποίο η πρόταση για τα πιλωτικά ε, ε, ομόλογα έργου για τις μεταφορές της επικοινωνίας και τις υποδομές ε, έχει ε, προταθεί και ε, για τον τρόπο με τον οποίο το χειριστήκατε. Επίσης εκτιμώ τις προσπάθειες για επίτευξη συμφωνίας για το αποκαλούμενο διπλό πακέτο που είναι ένα βασικό στοιχείο για τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ενίσχυση της οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας. Είναι ένα πρώτο βήμα για την εφαρμογή των σημαντικών στοιχείων του, του Δημοσιονομικού Συμφώνου. Γι' αυτό και ελπίζω ε, ότι το, ε, το Κοινοβούλιο υπό την Κυπριακή Προεδρία θα μπορέσει να φτάσει σε συμφωνία ε, πριν το τέλος του τρέχοντος έτους. Επίσης, συνεργασία για την φόρο για τις δημοσιονομικές για τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές ε, και ελπίζουμε ότι θα υπάρξει συμφωνία για τα παράγωγα μέσα στο χρόνο. Επίσης έχουν γίνει πρόοδοι όσον αφορά τις ε, εταιρείε αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Δεν έχουμε βρει βέβαια απόλυτη ομοφωνία ανάμεσα στα κράτη-μέλη, αλλά θα ήθελα να καλωσορίσω την απόφαση για αυξημένη συνεργασία για όλα τα κάτι που θέλουν να προσχωρήσουν σε αυτή την πρωτοβουλία. Πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή εξάλλου και πάλι είδαμε στους τελευταίους μήνες και εβδομάδες τόσο στη ΣΥΠΑ όσο και στην Ευρώπη μάλιστα και με μερικά από τα μεγαλύτερα τραπεζικά ε, ιδρύματα ότι οι λόγοι που οδήγησαν στην κρίση δεν έχουν εκκριζωθεί απόλυτα από τον τομέα. Έχουμε δηλαδή ε, δίσταχτη εμπορία ε, και κερδοσκοπία και αυτά θα πρέπει να εκκριζωθούν μια και παντός. Και θα πρέπει ο τραπεζικός τομέας να δεχτεί να δώσει ένα δίκαιο μερίδιο και στην κοινωνία. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρωθυπουργέ, αξιότιμοι κύριοι βουλευτέ, σε σχέση με τι πολύ δύσκολε διαπραγματεύσει για την προτινόμενη οδηγία για την επάρκεια στην ενέργεια, η συμφωνία που εξευρέθη από του συνομοθέτε στην πρώτη ανάγνωση ήταν ένα βασικό ε, ένα βασικό βήμα για την εξοικονόμηση 20% μέχρι το 2020. Έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε περίπου τα 2 τρίτα των συνολικών εξοικονομήσεων ενέργειας ε, από την πρόταση, σε σχέση με την αρχική πρόταση της Κομισιόν. Ε, βέβαια θα πρέπει να γίνει περισσότερη δουλειά για την επίτευξη των στόχων του 2020. Ε, επίσης πολύ σημαντική συμφωνία του περιαγωγής 3 που θα ωφελήσει τους πολίτες και τους καταναλωτές. Έχει αρχίσει να ισχύει από πρώτης ε, ε, εβδόμου. Έτσι κάναμε ένα σημαντικό βήμα για να προστατέψουμε τους καταναλωτές από ε, ε, σοκαριστικούς λογαριασμούς. Επίσης καλωσορίζουμε τη συμφωνία που επετέφθη για τη μεταρρύθμιση του συστήματος τυποποίησης που θα επιτρέψει πιο αποτελεσματικά πρότυπα στην Ευρώπη. Έχουμε επίσης επισφαλή κεφάλαια, ε, καθώς και τα ταμεία για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, καθώς και την επίλυση των διαφορών. Ε, πολύ σύντομα θα επιτευχθεί και εκεί συμφωνία. Και για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων έχει σημειωθεί πολύ σημαντική πρόοδος. Επίσης θα πρέπει να συζητήσουμε για το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα βριστεχνίας Για δεκαετίες συζητιέται. Εκεί βρέθη συμφω... Συμφω... συμβιβαστική λύση ανάμεσα στα συμμετέχοντα Όμω, Όμως δυστυχώς έρχεται με τίμημα την διαγραφή σημαντικών στοιχείων τη αρχική πρόταση τη Κομισιόν. Ενώ αναγνωρίζονται οι μεγάλες προσπάθειες ε, της Δανική για αυτό το σημαντικό θέμα και σα ευχαριστώ για αυτή την προσπάθεια, η Κομισιόν επιφυλάσσεται όσον αφορά τη θέση της και αυτή την επιφύλαξη την έχουμε καταστήσει σαφή στους επικεφαλής κατών και κυβερνήσεων στο Συμβούλιο. Χρειάζεται αξιολόγηση ανάμεσα στα τρία θεσμικά όργανα και είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε μαζί σας γι' αυτό. Κύριε Πρόεδρε, Το Ευρωπα... Επίσης προωθήθηκε το θέμα του πολυμερούς ε, ε, της ε, του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Το διαπραγματευτικό κοιτίο προετοιμάστηκε κατά τη διάρκεια της Δανέζικης Προεδρίας με στόχο να επιτευχθεί η συμφωνία μέχρι τα τέλη του 2012. Ως προς αυτό θα ήθελα να επαναλάβω ότι η Κομισιόν γνωρίζει πάρα πολύ καλά την έκκλησή σας για πλήρη σεβασμό των αρμοδιοτήτων κάθε θεσμικού οργάνου. Η Κομισιόν μάλιστα επέμεινε εντόνω σε αυτό το θέμα κατά τη διάρκεια τη προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και κατά τη διάρκεια τη έγκριση των συμπερασμάτων του. Η συζήτηση για το ΠΔΠ τώρα θα μπει στην τελική ευθεία. Θα πρέπει να υπογραμμίσω πω η Κομισιόν θεωρεί πω ακόμα λείπουν σημαντικά στοιχεία από το διαπραγματευτικό κοιτίο και δεν δίνονται απαντήσει σε κάποιου τομεί κατά τη γνώμη μα. Ενώ αναγνωρίζουμε την πολύ σοβαρή εργασία που έχει γίνει μέχρι στιγμή, η Κομισιόν θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τι προτάσει τη υπό την επερχόμενη Προεδρία και, και είναι σαφές τώρα ότι ο, δημοσιο... ο προϋπολογισμός της Ένωσης είναι ένα σημαντικό εργαλείο για να επιτευχθεί η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση μέχρι τις επενδύσεις της βιώσιμης ανάπτυξης των θέσεων απασχόλησης. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο που έχουν συνεργαστεί μαζί μας στενά. Ε, υπήρξε μια μακρά διαδικασία διαπραγματεύσεων και η τελική έγκριση πριν από το τέλος του έτους αυτού του ΠΔΠ θα είναι πολύ σημαντική. Γι' αυτό, επ' αυτού ελπίζω εντόνως ότι το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο με τη στήριξη της Κομισιόν θα καταφέρουν να φτάσουν σε αυτή τη συμφωνία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται να στείλει ένα μήνυμα ότι μέχρι το τέλος αυτής της δεκαετίας θα έχει έναν ισχυρό ε, προπολογισμό για την άπτυξη και τη συνοχή και να δείξει πως είναι σε θέση να λάβει αποφάσεις δύσκολες σε δύσκολους καιρούς. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ και αξιότιμοι κύριοι βουλευτέ, στον τομέα τη δικαιοσύνη και των εσωτερικών υποθέσεων έχει υπάρξει επίση πρόοδο, Δουβλίνο 2 και η οδηγία περί όρων ε, υποδοχή. Ε, έχει προχωρήσει και το θέμα του οδηγία για, για το άσυλο, αλλά και η μεταρρύθμιση των θεωρήσεων. Ωστόσο, δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο για ένα σημαντικό φάκελο, δηλαδή το θέμα της νομικής βάσης και της φύσης του μηχανισμού αξιολόγησης Σέγγεν, Όλοι γνωρίζουμε πόσο ευαίσθητο είναι αυτό το θέμα και όσον αφορά την Κομισιόν θέλουμε λύσεις που να μπορούν να λειτουργήσουν. Γι' αυτό πιστεύουμε αποκοινούμε το Κοινοβούλιο ότι χρειάζεται ένας μηχανισμός αξιολόγησης έγκαιων με ισχυρή ευρωπαϊκή διάσταση. Είμαστε πεπισμένοι πως ένα μοντέλο διακυβερνητικό δεν θα αποδώσει όσον αφορά την εντολή του Συμβουλίου του Μαρτίου 2011. Όλα αυτά είναι πολύ περιοριστικά στην πράξη. Και τέλος, με την ε, Λισαβόνα, η ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων είναι μια πραγματική ε, ανησυχία. Δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτό λοιπόν ως τελικό αποτέλεσμα και θα δουλέψουμε για μια καλύτερη λύση. Mr. President, Prime Minister, Πρόεδρε, ε, Πρωθυπουργέ, κύριοι Ευρωβουλευτές, εξωτερική διάσταση τώρα. Ε, πρέπει πάντοτε να συνδυάζεται αυτό με την ευρύτερη διάσταση του ρόλου της Ευρώπης στον κόσμο. Αυτό θα πρέπει να γίνει με, απορο... με αποφάσεις και προετοιμασία για το ε, Europe Sin εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μείνει προσιλωμένη και επικοδομητική κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και οι θέσει μα είχαν αντίκτυπο στη συζήτηση. Θα ήθελα να καλωσορίσω την πολύ καλή συνεργασία ανάμεσα στην Κομισιόν και την ε, Προεδρία της Δανίας. Και οι δύο, και, και η ε, Πρωθυπουργός ε, Σμίτ αλλά και εγώ ήμασταν παρόντες στη ορίο θα πρέπει να σας πω ότι αυτή η διάσκεψη δεν θα έχει πετύχει αυτό το σημαντικό αποτέλεσμα. Πράσινη ανάπτυξη πλέον ρητά και επισήμως είναι αποδεκτή από τη διεθνή κοινότητα ως απαραίτητο τμήμα της, βιώσιμης, της ατζέντας βιώσιμης ανάπτυξης. Σημαντική πρόοδος έχει επιτευχθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι μηνών της Δανέζικης Προεδρίας και θέλω να ευχαριστήσω ακόμη μια φορά για την πολύ καλή συνεργασία. Αλλά γνωρίζουμε πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση, πόσο ακόμα, πόσο ακόμα πράγματα πρέπει να πετύχουμε. Ε, ελπίζω λοιπόν ότι θα έχουμε τη συνεργασία όλων για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτές τις προκλήσεις. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα ο κύριος Κάρινς, ε, εκπρόσωπος του ΕΛΚ, έχει τον λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρωθυπουργέ, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής. Υπό συνθήκες ε, οικονομικής κρίσης η τάση, η συνήθιση είναι να επικεντρώνουμε τις προσπάθειές μας ε, ούτως ώστε να μπορέσουμε να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο και όλα τα άλλα να τα παραμελούμε. Και όλοι γνωρίζουμε ότι το τελευταίο εξάμεινο και όχι μόνο κατά αυτή την περίοδο ε, αυτό το οποίο βασικά θέλαμε και αυτό το οποίο συνεχώς έβγαινε στον τύπο ήταν η χρηματοπιστωτική κρίση. Η Προεδρία της ε, Δανίας επομένως ε, έπρεπε να ασχοληθεί με το θέμα αυτό και τα άλλα να παραμεληθούν. Πάρα πολύ σημαντικό το θέμα της κρίσης φυσικά, όμως θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι με θάρρος η Προεδρία ασχολήθηκε και με άλλα πολύ σημαντικά προβλήματα και αναζήτησε και για τα άλλα προβλήματα κάποιες λύσεις. Όχι, δεν θέλω τώρα να επαναλάβω αυτό το οποίο είπε ο πρόεδρος Επιτροπής. Αυτό το οποίο θέλω να σας τονίσω είναι ε, το τι έγινε με την ενεργειακή πολιτική. Διότι είναι θέμα πάρα πολύ σημαντικό για το μέλλον και επίσης θα πρέπει να συγκροτηθεί μια κοινή ενεργειακή πολιτική. Έτσι να μπορούμε να έχουμε ασφαλή προμήθεια της ε, ενεργείας, να έχουμε πιο καθαρή ενέργεια και επίσης κάτι το οποίο είναι σημαντικό να μην εξαρτώμεθα από το εξωτερικό για τα, τις εισαγωγές μας. Οπότε και η Δανέζικη Προεδρία ασχολήθηκε με το θέμα αυτό. Το Δεκέμβριο θα ψηφίσουμε σχετικά θα δούμε τι θα γίνει με τις ε, συμφωνίες εισαγωγής από τρίτες χώρες. Η Δανέσκη Προεδρία ε, εδώ είχε να αντιμετωπίσει τις αντιρρήσεις κάποιων κρατών μελών που δεν συμφωνούσαν με την σχετική νομοθεσία. Όμως τελικά κατάφερε η Δανέσκη Προεδρία να κλείσει ένας ε, συμβιβασμός. Αυτό και θα ψηφίσουμε τον Δεκέμβριο. Αυτό σίγουρα είναι μια πρόοδος ένα βήμα προς το να αποκτήσουμε μια κοινή πολιτική ενέργεια. Οπότε θα πρέπει και να ευχαριστήσουμε την ε, Δανειστική Προεδρία. Ε, ασχολήθηκε και με την κρίση, αλλά και με άλλα θέματα. Ευχαριστώ κύριε Κάριν, και τώρα για τους σοσιαλιστές ο κύριος Φόμποντα. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρωθυπουργέ, καταρχήν ευχαριστώ την Προεδρία και ευχαριστώ για τον κατάλογο τον οποίο διαβάσατε σήμερα το πρωί για όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της Δανικής Προεδρίας και πρέπει να αναγνωρίσω ότι είναι ένας εντυπωσιακός κατάλογος. Βεβαίως η Προεδρία αυτή σκιάστηκε από δύο παράγοντες στην οικονομική κρίση και χαίρομαι διότι στο τελευταίο Συμβούλιο Κορυφής μπόρεσαν να γίνουν κάποια θετικά βήματα προς την ανάπτυξη που είναι είναι απαραίτητο στοιχείο για να αντεπεξέλθουμε τις κρίσεις και του Συμβουλίου. Αναφέρατε το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρασιτεχνίας. Ε, το Κοινοβούλιο όμως μάχεται χρόνια για το δίπλωμα αυτό για να μπορέσει να επιλύσει το πρόβλημα των, των επιφυλάξεων πορών χωρών ε, και μπορέσαμε τελικά να καταλήξουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα αλλά βλέπω ότι Μεγάλη Βρετανία η οποία πάντοτε πιέζει διότι έχουμε τρία, τρεις έδρες για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνει τρεις έδρες για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας βλέπετε εδώ τι γίνεται με τις κυβερνήσεις επίσης για τον προπολογισμό και εκεί έβαλε το χέρι του το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και πρέπει να σας πω ότι ε, ε, ο κύριος Βανορόμποη ε, είπε πολύ σωστά ότι το Συμβούλιο πρέπει να ασχολείται με τα του οίκου του και να μην εμπλέκεται σε θέματα τα οποία πρέπει να γίνονται από κοινού και να αποφασίζονται όπως η νομοθεσία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίση, θα ήθελα να τονίσω την οδηγία για την ενεργειακή αποτελεσματικότητα. Πρόκειται για μια κατεύθυνση όπως είπε ο κύριο Τούρμες και η κυρία Μπρίτα Τόμσον τα προώθησαν. Είμαστε ευγνώμονες προς αυτούς και πάλι όμω ορισμένα κράτη εμπόδισαν να γίνει ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός. Και ελπίζω ότι με την βοήθειά σα σαν εκπρόσωπο τη Δανία ότι θα μπορέσει να γίνει αυτή η στροφή στην ενέργεια να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις εκατοντάδες χιλιάδες θέσεων εργασίας. Ψάχνουμε πού πήγε η δουλειά, πού πήγε η απασχόληση. Εάν όμως εστιαστούμε στο πρασίνισμα της οικονομίας θα δημιουργηθούν πολλές θέσεις στην Ευρώπη και θα μειωθεί και η εξάρτηση από τις εισαγωγές αερίου και πετρελαίου. Αυτά επιτέχθησαν και ελπίζω ότι ορισμένες χώρες οι οποίες αντεστάθησαν μέχρι τώρα θα μπορέσουν να συμφωνήσουν ότι στο μέλλον χρειαζόμαστε ενεργειακή αποτελεσματικότητα. Και τέλος όσον αφορά την επιλογή σας κύριε Πρωθυπουργέ ε, για τον Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων θέλω να σας συγχαρώ διότι εργάστηκε ο εκπρόσωπός σας ε, εξαιρετικά μας έδειξε πώς μπορεί κανείς να ε, λειτουργεί και για την Ευρώπη Ευρώπη και να προασπίζει τα συμφέροντα της χώρας του Γι' αυτό και σας ευχαριστώ όλους για την εργασία και τη συνεργασία σας. Ευχαριστώ. Κύριε Σβόμποντα, τώρα για τους φιλελεύθερους ο κύριος ε, Γκραφ Λάμπσδορφ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρία Πρωθυπουργέ. Ακούσαμε ότι το ευρωπαϊκό οικοδόμημα βασίζεται στα τουβλάκια της αλληλεγγύης, αλλά πρέπει τα, οι βάσεις να είναι ε, ισχυρές και γι' αυτό εάν θέλει κανείς να συνδυάσει την ασφάλεια και τη σταθερότητα με την αλληλεγγύη θα πρέπει να έχετε μιλήσει περισσότερο για την σταθερότητα πώς μπορούμε να ελέγξουμε καλύτερα την οικονομική κρίση. Ε, είπατε πολύ σωστά ότι στο Του pac μπορέσαμε, στο, στο διπλό πακέτο μπορέσαμε να προωθήσουμε θέματα τα οποία μας απασχολούν και η απόφαση του Σαββατοκύριακου στο Συμβούλιο αφήνει ανοιχτά πολλά θέματα. Ο κύριος Φόμποντα αναφέρθηκε στο σύμφωνο ανάπτυξης, είναι κάτι το οποίο τον ενδιαφέρει πολύ. Μίλησε για 50 έως 55 δισεκατομμύρια τα οποία πρέπει ε, να διατεθούν αλλά και ο Επίτροπος Χάν δεν ξέρει από πού θα προέλθουν. Άρα δεν ξέρω αν υπάρχει τόση σταθερότητα. Όντως θα πρέπει να προχωρούμε από κοινού. Ναι, θέλουμε να δημιουργήσουμε απασχόληση θέλουμε το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας αλλά είναι ανόητο όπως σωστά είπε ο κύριος Βόμποντα να έχουμε ένα όργανο με, τρία, με τρεις έδρες το Λονδίνο, το Παρίσι και το Μόναχο σε ένα τόσο σημαντικό καινοτόμο θέμα δεν είναι δυνατόν να καταλήγουμε σε αυτή την απόφαση επίσης το άρθρο 127 ε, παράγραφος 6 προβλέπει τώρα ότι θα υπάρξει μία νέα αρχή εποπτείας των τραπεζών στην Ευρώπη αλλά νόμιζα ότι είχαμε μία αν έχουμε τώρα δύο έδρες θα υπάρχουν ε, ε, δύο ε, ε, ε, ε, εποπτείες και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να στηρίξει τέτοιες προσπάθειες αντιφατικές όταν προσπαθούμε να εξοικονομήσουμε πόρους. Κατά τα άλλα όντως προχωρήσαμε, δεν αναφέρθηκα στο Σέγγεν που ήταν ένα θαύμα της Προεδρίας σας αλλά η συνεργασία με τη Σερβία και το Μαυροβούνιο όντως ήταν πολύ επικοδομητική. Ευχαριστώ τώρα για τους πράσινους ο κύριο κύριος Κον Μπεντίτ. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε, μάλλον ας σκεφτούμε ότι κάποια στιγμή έχουμε μια Προεδρία, έναν Πρόεδρο της Επιτροπής, ο οποίος έρχεται εδώ μετά από το ένα εξάμεινο από μια Προεδρία και μας λέει «Ε, τα ξέρετε, ξέρετε τι κάναμε. Κάναμε πολλά. Α, όντως, τα κάναμε με δυναμισμό, όμως τώρα, για να δούμε πού φρακάρισε το θέμα γιατί εδώ μαζί θα πρέπει να γνωρίσουμε δεν είναι το θέμα ότι δεν είχατε κάποιο όραμα αλλά δεν καταλαβαίνουμε πάντοτε γιατί δεν μπορέσατε να το υλοποιήσετε το όραμά σα γιατί μα μιλήσατε για εκείνη την οδηγία όσον αφορά την αποτελεσματική χρήση τη ενέργεια, αλλά α μην γελιόμαστε ήταν δύο χώρε οι οποίε φρέναραν αυτή την, την υπόθεση ε, ο Γερμανο, υπουργό κ. Λάμστορφ και η Πολωνία. Άρα θα πρέπει κάποια στιγμή να συζητήσουμε πω θα απεμπλακεί η ευρωπαϊκή υπόθεση. Γιατί τι γίνεται, να, όπως, ε, όπως το σινεμά, λέμε, α, ωραία, συνεργαστήκαμε και, και πολύ καλά γνωρίζουμε ότι οι αποφάσεις που λαμβάνουμε δεν είναι στο ύψος των περιστάσεων. Η οδηγία για την ενέργεια έχει καλώς, όμως όλοι γνωρίζουμε ότι δεν αρκεί. Και δεν φταίτε εσείς. Φταίει ο τρόπος λειτουργίας της Ευρώπης. Μιλήσαμε για την ευρεσιτεχνία. Ε, είναι παράλογο. Θα πρέπει κάποια στιγμή να το καταφέρουμε, θα πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος το πρόβλημα. Δεν είναι αυτά, που εδώ λέμε, είναι αυτό το τι μπορεί να καταλάβει η κοινή γνώμη. Και όταν υπάρχει αυτή η αντίφαση μεταξύ του κυρίου Κάμερον, ο οποίο υπαγορεύει όλο τον κόσμο τι πρέπει να κάνει, αλλά από την άλλη μεριά φρενάρει την Ευρώπη, ε, θα πρέπει ο κόσμο, η κοινή γνώμη, α πούμε για τι ευρεσιτεχνίε, να να ξέρει τι γίνεται. Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα όπως το Σέγγεν. Το Σέγγεν είναι ξεκάθαρη περίπτωση. Εάν ε, η υπόθεση άνοιγμα κλείσιμο συνόρων ξαναγίνει εθνική υπόθεση, αυτό θα είναι η ταφόπλακα στην, ε, στο, ευρωπαϊκό όραμα και ε, τελικά την ευθύνη τη φέρνουν οι Υπουργοί Εσωτερικών, μας τα πράγματα με το όνομά τους για να καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται πραγματικά. Και μας είπατε επίσης και για την ένταξη του Μαυροβουνίου και της Σερβίας. Σύμφωνοι. Αλλά ακόμη μια φορά, ακόμη μια φορά, ξεχνάμε τι έγινε στο Σαράγεβο, ξεχνάμε τι έγινε στην Βοσνία. Την ξεχνάμε τη Βοσνία γιατί σήμερα η μόνη χώρα που δεν έχει ευρωπαϊκή προοπτική είναι εκείνη που έπεσε θύμα του, του, του εθνικισμού στα Βαλκάνια. Η Βοσνία. Νομίζω ότι ε, λέτε απλώς ωραία λόγια ε, ε, αλλά εάν δεν βρείτε μια λύση που να καλύπτει και την Βοσνία εγώ θα συνεχίσω να θεωρώ τα πράγματα είναι άσχημη θα έχω Ευχαριστώ τώρα για τους Ευρωπαίους συντηρητικούς ο κύριος Κάλαχαν Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε Δύο την ε, κράτησα από τα όσα άκουσα σήμερα το πρωί. Πρώτα πρώτα θα πρέπει σε, να πω χρόνια πολλά στο Γενικό Γραμματέα μας. Είμαι σίγουρος ότι είναι ενθουσιασμένο με όλα αυτά τα συγκλονιστικά που ακούει τώρα που γιορτάζει. Αλλά δεύτερο και σημαντικό είναι το να ευχαριστήσω την Δανέζικη Προεδρία. Τους συνεργάτες των Υπουργών, τους Υπουργούς βέβαια, όλοι αυτοί που ασχολήθηκαν με την Προεδρία το τελευταίο εξάμεινο. Βεβαίως, και οι σοσιαλιστές και εγώ σε συντηρητικός ε, σε κάποια θέματα διαφωνούμε Παρ' αυτά όμως θα πρέπει τη χαρακτηριστική σας δανέζικη πρακτικότητα και αποτελεσματικότητα ε, να την ε, επενέσω για όσα κάνετε τελευταία εξάμεινο και βεβαίως θα πρέπει να σας συγχαρούμε γιατί θάψατε τον φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Αυτό το οποίο θα, θα, θα χτυπούσε πολλά κέντρα συναλλαγών και πάρα πολλούς συναλλαζομένους αποταμιευτές. Επίσης ε, θα πρέπει να δούμε τι έγινε, την οδηγία για τους εργαζόμενους. Ε, αυτό το οποίο θα, θα δυσκόλευε πάρα πολύ το να βρουν θέση, πάρα πολλές, θέση εργασίας πάρα πολλές γυναίκες και κάνει τις εργασίες επίσης ε, όσον αφορά τα μέτρα λιτότητα στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, τα μέτρα συγκράτηση δημοσιονομικών δαπανών δηλαδή που επιβάλλατε, γιατί θα μπορούσατε ε, στους σοσιαλιστέ, του άλλους, πάρα πολλά να του πείτε, να τους, να τους, να να, να, να γίνεται παράδειγμα προ μίμηση, ε, του σοσιαλιστέ που κάνουν πειράματα στην εξουσία. Τώρα, όσον αφορά την, τον μηχανισμό αξιολόγηση του Σέγγεν, θα πρέπει να σα πω ότι καταλαβαίνω Καταλαβαίνω ότι, περνάτε γιατί έγινε η αλλαγή της ε, νομικής βάσης ομόφωνα στο Συμβούλιο και ο κύριος Ντόλ μας το, μας το ξαναείπε ότι αυτό το κάνανε κυρίως, κυρίως οι ηγέτες του ΕΛΚ. Επομένως ε, δεν θα πρέπει να πυροβολούμε τον, ε, τον ταχυδρόμο είπαμε επίσης, η Ιδανική Προεδρία επίσης είχε εργαστεί συνεργασία, καλή σχέση με το Κοινοβούλιο και βεβαίω και ο κ. Ρόιμαν, ο υπουργό σα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, ο οποίο ερχόταν και ξαναρχόταν εδώ πέρα και ε, τα, τα άκουγε, υφίστατο πάρα πολλέ ε, επικρίσει, αλλά όλα αυτά τα υπέστη ε, στοικά και επομένω το μέλλον ξανοίγεται μπροστά του ρόδινο. Οπότε θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι πάρα πολύ καλά τα πήγαμε και φυσικά η Δανέζικη Προεδρία, επομένω μόνο θετικά σχόλια μπορεί να αποσπάσει. Ευχαριστώ κύριε Κάλαχαν <clears throat> και τώρα για την Ηνωμένη Αριστερά το λόγο έχει ο κύριος Ζόντεργκαρτ. Ευχαριστώ. Πέρσι η Δανέζικη Προεδρία μας είπε ότι η επιστροφή της ανάπτυξης αλλά και ψηλός ρυθμός απασχόλησης θα πρέπει να εξασφαλιστούν και βραχυπρόθεσμα και μακρόπνοα. Και να δούμε τώρα εάν έκαναν αυτά τα οποία είπαν γιατί βραχυπρόθεσμα δεν μπορούμε να πούμε ότι τήρησαν την υπόσχεσή τους η, ε, η, της κυβέρνησης της Δανίας. Είδαμε τι έγινε με τα στοιχεία για την ανεργία. Πρόκειται για μια τραγωδία γιατί ποτέ, ποτέ στην Ευρώπη δεν είχαμε τόσους ανέργους. Ε, πρόκειται για μια τραγωδία. Πρόκειται για μια τραγωδία. Και αυτό γιατί έγινε λόγω των μέτρων που έλαβε η Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω των μέτρων που ε, την πρώτη μέρα τη προεδρία τη υπεστήριξε η Δανέζικη Προεδρία. Τι έγινε στην Δανία, στην Ιρλανδία. ακριβώ, λόγω της κρίσης θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλες περικοπέ. Τόσο μεγάλε που η Ιρλανδία ε, έπρεπε να κόψει τα δύο τρίτα του προπολισμού για την παιδεία. Με τίποτα επομένω δεν μπορούν να καλυφθούν οι συνέπειε ε, από αυτές όλες τις περικοπές. Έχουμε πάνω από 25 εκατομμύρια ανέργους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο προχωρεί σε ένα πρόγραμμα για την απασχόληση που δεν έχει όμως συγκεκριμένους στόχους όσον αφορά το πώς θα συγκρατηθεί το φαινόμενο αυτό της ανεργίας. Στην αρχή ε, της Δανεικής Προεδρίας είχα λάβει το λόγο, είχα μιλήσει και είπα ότι οι Ευρωπαίοι δεν αντέχουν άλλες περικοπές. Θέλουν, χρειάζονται περισσότερες θέσεις απασχόλησης, χρειάζονται περισσότερο κράτος ευημερίας. Η Δανεική Προεδρία ήταν μέρος της λύσης ή μέρος του προβλήματος. Δυστυχώς θα πρέπει να καταλήξουμε εμείς ότι όσον αφορά την απασχόληση, η Δανειακή Προεδρία δεν ήταν το τμήμα της λύσης. Τον λόγο τώρα ε, για την ΕΦΤΕ ο κύριος Μέσερ Σμιτ. Τα καταφέρατε. Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, κανείς ποτέ δεν κατάφερε να ξεπουλήσει τόσο πολλά και παρόλα αυτά δεν πετύχει τίποτα γιατί δεχτήκατε το μέτρο των χρηματοπιστωτικών ε, νομοθετημάτων ε, για το Σέγγεν επίσης προχωρήσατε ε, και στην γεωργική πολιτική κάνατε ό,τι μπορούσατε και επίσης ματαιώσατε τα δημοψηφίσματα και επίσης προσπαθήσατε κάτι να κάνετε και για την, ε, ε, το Δήμο της Τελικά ε, το love story έγινε, έγινε σαπουνόπερα. Θα μπορούσατε να πετύχετε πολλά, αλλά δεν καταφέρατε. Και ουσιαστικά αυτό το οποίο κάνατε ήταν το, το, το, το ευρωπαϊκό τιτανικό να τον βυθίσετε και αυτή τη στιγμή δεν είναι πάνω στο παγόβουνο ιτανικό, είναι στο βυθό τη θάλασσα. Και δεν νομίζουμε ότι μπορεί εύκολα να γίνει ναυαγιέρεση, γιατί κάνατε τη μία συνέντευξη μετά την άλλη, αλλά τελικά βάλατε την ταφόπετρα στο, στο, στην ευρωπαϊκή οικονομία οπότε σας ξεκαθαρίζουμε κάτι το οποίο ελπίζω να καταλάβετε ντροπή, ντροπή σας διότι άκουσα ότι πάρα πολλοί εξεπλάγησαν που δεν είχατε όραμα ως Προεδρία ακόμα και οι Γάλλοι σοσιαλιστές φίλοι σας εξεπλάγησαν όμως, όμως τελικά δεν πρόκειται για μια συνήθεια Προεδρία. Ήταν σαν κανείς να, κάνει, να περνάει μια συνέντευξη για να πιάσει δουλειά. Αλλά παρακράτησε πολύ αυτή η συνέντευξη. Αλλά καλά, πάντως εσείς δεν θα ξαναβγείτε πρωθυπουργό, αν και φαντάζομαι ότι θέλετε να γίνετε πρόεδρος της Κομισιόν ή να γίνετε μόνιμη πρόεδρος του Συμβουλίου, τόσο ώστε να βλέπετε και να ξαναβλέπετε του φιλαράκου σα εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, κύριε Μπαρόσο και ο κύριο Βανεροπόη θα πρέπει να ανησυχούν γιατί υπάρχει τώρα εδώ αυτή η κυρία η οποία θα κάνει ό,τι να είναι, ό,τι μπορεί για να πετύχει αυτά τα οποία θέλει. Και το, το είδαμε αυτό επανειλημμένα σε αυτό το εξάμεινο. Οπότε ε, νομίζω ότι οι περισσότεροι Δανείοι θα συμφωνούν μαζί μου. Παρακαλώ, κυρία Τόνι Σμιθ, ξανά ελάτε εδώ, ελάτε εδώ και αφήστε με εσεί <clears throat> Κυρίες και κύριοι, λοιπόν, ηρεμήσατε, εντάξει. Ο κύριος, προς τον κύριο Μέσερσμιτ θέλω να το ρωτήσω. Ο κύριος Ρόντε, ο συνάδελφός σας, θέλει να θέσει μία ερώτηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Το παράκανε ο κύριος Μέσης, ακόμα και για τα δικά του δεδομένα. Ίσως για όλα αυτά που έλεγε, ιδίως όταν λέγει εντροπή, θα πρέπει να κοιτάει κανένα καθρέφτη. Τι να σας πω. στόματος κόρακος κρά. Λοιπόν, ε, τι κάνετε, ανησυχείτε τόσο πολύ για την Ευρωπαϊκή Τεχνία. Μα, κύριε Μέσεσμιτ, εσείς θέλατε στη Δανία να γίνει δημοψήφισμα για τις ε, ευρωπαϊκές ε, ευρεσιτεχνίες τα διπλώματα και τώρα μας λέτε δεν θέλετε να υπάρξει ευρεσιτεχνία και τι μας λέτε, για, μας λέτε για όλους εκείνους, για όλες τις εταιρείες που επί 30 χρόνια ζητούν να θεσπιστεί ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ευρωπαϊκό ούτως ώστε να είναι φτηνότερο οι ευρωπαϊκές εταιρείες να, να μπορούν να το έχουν αυτό και να έχουν και ανταγωνιστικότητα. Μέσα σημαίνει Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την ερώτηση. Πρώτα-πρώτα όσον αφορά το δημοψήφισμα ή τα δημοψηφίσματα. Εγώ πιστεύω στα δημοψηφίσματα. Διαφωνήσαμε όσον αφορά το τελευταίο δημοψήφισμα. Επομένω, δεν σα φαίνεται τόσο περίεργο το ότι αφού τώρα μα δίνει τη δυνατότητα το Σύνταγμα να λέμε ότι χρειάζεται για την Ευρωπαϊκή Ευρεσιτεχνία να γίνει δημοψήφισμα. Και αυτό το οποίο μα ανησυχεί είναι το, το, το, το κατά πόσον ε, κανένας μπορεί να κάνει forum shopping, να πηγαίνει όπου τον βολεύει η ρύθμιση και να μπλέκονται τα εθνικά δικαστήρια, να μην μπορεί κανείς να προσφύγει σε κάποια κεντρική ευρωπαϊκή αρχή. Ε, αυτό είναι πρόβλημα. Ε, και τελικά, ποιο, δεν ξέρω, εσείς θέλετε να, ε, να ωφελήσετε τι πολυεθνικέ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σήμερα συζητάμε για το πρώτο εξάμεινο 2012. Το 2012 έχει χαρακτηριστεί από την αποτυχία της Ευρώπης, από την απώλεια εμπιστοσύνη των πολιτών στο ευρωπαϊκό όνειρο, το οποίο έχει αποτύχει. Μία ολόκληρη σειρά από χώρες του Νότου είναι στα πρόθυρα της ε, κατάρρευσης. Ε, στα κράτη-μέλη ε, ε, λέει, λατούνται τα ταμεία δήθεν ε, χα, προς χάρη αλληλεγγύης. Αν συνεχιστεί αυτή η τάση, ε, διαρωτάται κανείς αν αύριο θα υπάρχουν όλες αυτές οι χώρες. Πολλές χώρες ζητούν την κατάργηση πια του ευρώ. Εγώ συμφωνώ, γιατί αν δεν ε, μπορεί να σταθεί το ευρώ δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Κύριος Βανέστερ Ρόι. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την, τους εκπροσώπους του Συμβουλίου και της Κομισιόν για τις προόδους που έχουν ε, επιτευχθεί, ιδιαίτερα η Συμφωνία για την Ενεργειακή Επάρκεια αλλά και για τις διάφορες δημοσιονομικές συμφωνίες. Επιπλέον υλοποιήσαμε σημαντικούς στόχους και σε άλλες και σε άλλους τομείς, ο συντονιστής του ΕΛΚΑ για τη ε, περιφερειακά θέματα, ε, συνειδητοποιώ ότι σε άλλους τομείς λείπουν οι ε, πρόοδοι. Εάν δεν φτάσουμε σε συμφωνία εντός του τέλος του έτους, ε, δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να εφαρμόσουμε τον κανονισμό για το ΠΔΠ. Φυσικά έχει υπάρξει πρόοδος όσον αφορά τον κανονισμό για τα διαρθρωτικά ταμεία. Η συναπόφαση του Κοινοβουλίου κάπως μπήκε εντός παρεθέσεως γιατί πολλές αποφάσεις αναβλήθηκαν για την ε, στιγμή της έγκρισης του ΠΔΠ. Ας δούμε λίγο το άρθρο 312 τη συνθήκη της Λισαβόνας ή το άρθρο 174-176. Ορίζεται εκεί μία θεσμική αρχιτεκτονική που θα πρέπει να, να θεωρηθεί ή να αποκατασταθεί. Δηλαδή ή θέλει το Συμβούλιο ολόκληρε το θέμα του δημοσιονομικού πλαισίου να πέσει και πάλι ε, υπό την αρχή της συναπόφασης. Εμείς θέλουμε να τηρηθεί η συνθήκη της Λισαβόνας. Μετά από την ψηφοφορία της 15ης ε, Ιουλίου με εντολή της Επιτροπής μας θέλουμε από κοινού να αντιμετωπίσουμε τα θέματα που μας είναι ιδιαίτερα προσφυλή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Βαλνίστελ Ρόι. Ο κύριος Κάλαχαν με συνεχάρη για τα γενέθλια και ε, συνεχάρη τον εορτάζοντα για την, ε, τα γενέθλια. Υπάρχει όμως και κάποιος άλλος ο οποίος πρέπει να συγχαρούμε σε αυτό το κοινοβούλιο ε, και έπρεπε να περιμένω να είναι εδώ. Πρόκειται για τον Τζέρσι Μπούζεκ που έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Τον συγχαίρω του εύχομαι ό,τι καλύτερο. Τζέρζι ήθελα να σε συγχαρούμε από τον Γενικό Γραμματέα γιατί ο Γενικός Γραμματέας και ο Πρόεδρος μέχρι τώρα είχαν μαζί τα γενέθλιά τους τώρα όμως δυστυχώς έχουν χωρίσει τύχες τους. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Γιόργενσεν. Ε, Ντάν, σε παρακαλώ το μικρόφωνο σου. Κύριε Πρόεδρε, η Ευρώπη αυτή τη στιγμή περνάει μια κρίση. Πάρα πολλέ χώρε βρίσκονται στο χείλο της κατάρρευσης και έχουμε τραγικούς ρυθμού ανάπτυξη και τραγικούς ρυθμού ανεργίας. Θα δούμε, πρέπει να δούμε κατά πόσο μπορούμε κάτι, κάτι, κάτι, να πετύχουμε συγκεκριμένο γιατί τα κράτη-μέλη θα πρέπει από κοινό να προχωρήσουν, να δημιουργήσουν πρόοδο, να ε, δημιουργήσουν κλίμα αισιοδοξία, κάτι το οποίο δεν είναι πάρα πολύ εύκολο, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι και είναι σημαντικό επίση το ότι η Δανέζικη Προεδρία τα πήγε πάρα πολύ καλά. Ήταν πετυχημένη. Δεν λέω ότι φρέναρε την, την κρίση και, όλα τα κανερόδινα φυσικά δεν είναι τίποτα τέτοιο. Όμως, όμως αυτό το εξάμεινο ελήφθησαν αποφάσεις που αποτελούν βήματα σημαντικά προς σωστή κατεύθυνση. Υπεύθυνη Ευρώπη, δυναμική Ευρώπη, πράσινη Ευρώπη, ασφαλής Ευρώπη. Όλα αυτά τα προχώρησε η Δανέζικη Προεδρία με συμβιβασμούς, ε, με διαβήματα τα οποία ήταν πάρα πολύ θετικά. Έχουμε πάνω από 20 εκατομμύρια ανέργους και κυρίως πάρα πολλούς νέους. Ε, είχαμε δηλαδή έκρηξη ρυθμών ανεργίας. Προσπάθησε κάτι να κάνει για την ανάπτυξη η Δανέσκη Προεδρία. Είχε και αυτό το, το, το πακέτο μέτρων ανάπτυξη, ε, το οποίο πρόκειται να δημιουργήσει δεκάδε χιλιάδε θέσει εργασία, το οποίο πρόκειται να ξαναβάλει ε, την, ανάπτυξη, την Ευρώπη στο δρόμο της ανάπτυξης χρειάζεται πάντως δημοσιονομική εξυγίανση. Πολλά άλλα πετύχατε, προχωρήσατε και την οδηγία για την ε, αποτελεσμένη χρήση της ενέργειας. Αυτό όπλας ε, οικολογικής ήταν πάρα πολύ φιλόδοξη νομοθεσία. Ε, ίσως πιο φιλόδοξο νομοθέτημα στον κόσμο που κάνατε, αλλά επίσης έτσι με την πολιτική ενώπιση του 2020 έχουμε δημιουργία θέσεων εργασίας. Έχουμε πάνω από 200. 250 επιτυχήμετρα, 250 αποφάσεις που ωφελούν τους Ευρωπαίους. Ε, αυτό είναι κάτι το οποίο ε, μπορεί να σας κάνει αισθάνεστε υπερήφανος και εμάς να κάνει υπερήφανος ε, και και εσάς επίσης αυτό πετύχατε. Το λόγο έχει τώρα ο συνάδελφος κύριος Γένς Ρόουντε για 1,5 λεπτό. Er σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι ε, έχουμε κάθε λόγο να σας συγχαρούμε για την Προεδρία σας. Επίσης, να ευχαριστήσουμε και τους συνεργάτες σας και τον ε, κύριο Νικολάη τον ε, Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, ο οποίος συνεργάστηκε πάρα πολύ με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ό,τι και να πρεσβεύει ο καθένας από εμά δεν μπορούμε παρά να αναγνωρίζουμε την συμβολή του κυρίου Υπουργού. Πάντως, Υπάρχουν και κάποια πράγματα τα οποία μας εξέπληξαν ε, από την Προεδρία. Ε, α, αυτό το οποίο τώρα για τον Κόνραντ Αντενάουρ στην ε, ομιλία σας στην αρχή της συνάντησής μας. Μιλήσατε επίσης και για την αλληλεγγύη. Μα δεν καταλαβαίνω. Τι έγινε την περασμένη εβδομάδα. Την περασμένη εβδομάδα αποστασιοποιηθήκατε από την κοινωτική αλληλεγγύη, από την υπόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είπατε ότι η Δανία δεν θέλει να στηρίξει άλλες χώρες ε, για το χρέος τους. Ήδη το είπατε και το κάνατε. Και ακυρώσατε και εκείνο το δημοψήφισμα στη χώρα μας, στη Δανία. Να, να σας πω ακριβώς πώς τα είπατε στην ομιλία σας. Ο, αρκετά πρόσφατα yeah, ε, ε, είχαμε κάποιους διεθνείς οργανισμούς που δεν κατάφεραν να κάνουν όλα αυτά τα οποία έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση του τελευταίου 6 μήνε. Έτσι είπατε. Μεγάλα, παχιά λόγια αυτά. Και νομίζω θα πρέπει να πείτε συγκεκριμένα ακριβώ τι κάνατε. Μα Ωραία, αφού λάβετε τόσο ωραίε αποφάσει, τόσο σημαντικέ αποφάσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε γιατί, γιατί δεν θέλετε δημοψήφισμα στη Δανία, αυτό θα πρέπει να, να κάνετε, κυρία Υπουργή Χρόνο ε, κυρίε και κύριοι συνάδελφοι. Επόμενη ομιλήτρια είναι η συνάδελφος κυρία Τούρουνεν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρωθυπουργέ. Ε, σας χαιρετίζω που ήρθατε πάλι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Την τελευταία φορά που είσαστε εδώ είχατε πει κάτι που με εξέπληξε, ότι καταλαβαίνετε όλους τους νέους οι οποίοι δεν έχουν κανένα μέλλον όπως έγινε με τη γενιά της δεκαετίας του 80. Το πρόβλημα όμως της ανεργίας δεν εξαλείφθηκε από τον Ιανουάριο. Αυτό όμως που είναι θετικό είναι ότι τώρα είμαστε πιο εστιασμένοι ε, στην ε, ανεργία από ότι πριν από έξι μήνες. Τότε μιλούσαμε για επιστροφές ενώ τώρα μιλάμε επίσης για τη δημιουργία ανάπτυξης και ε, απασχόλησης. Χρειάζονται όμως εχέγγυα. Δεν ε, πρέπει να συγχαρούμε μόνο την Δανική Προεδρία αλλά συνέβαλε στην απόφαση αυτή. Σας ευχαριστώ λοιπόν και εφόσον τελείωσε ο χρόνος μου πρέπει να σας πω ότι περάσαμε τις εξετάσεις μας επιτυχώς ε, σαν χώρα στην Προεδρία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Δανία ανέλαβε την Προεδρία σε μια δύσκολη πηγή, περίοδο διότι συζητήσαμε για το Δημοσιονομικό Σύμφωνο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ε, αντί να μιλάμε για την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς, της μείωσης των επιδοτήσεων και πραγματικής ανάπτυξης. Οι συνθήκες ήταν δύσκολες και θέλω να ευχαριστήσω τον ε, Υπουργό Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων τον Νικολάη Μπάμεν ο οποίος ε, ήταν στο Κοινοβούλιο και ε, ε, ενέπλεξε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις διεργασίες. Τον ευχαριστώ για αυτό και θέλω να τον ευχαριστήσω επίσης για την βοήθεια του στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ε, όσον αφορά τα επικίνδυνα χημικά πρέπει να πω ότι είμαι λίγο απογοητευμένος γιατί είπατε ότι θέλετε να αναθεωρήσετε ε, και την ε, πολιτική αλίας αλλά και αυτό με απογοήτευσε γιατί ανεκάλυψα ότι δεν υπάρχει ένα βιώσιμο σχέδιο και εκπλήσω μου ότι ένα τέτοιο σχέδιο καταρτίστηκε κατά την Δανική Προεδρία αλλά πρέπει να πω ότι η Προεδρία ήταν πολύ επαγγελματική. Καλώς το βήμα τον συνάδελφο κύριο Αντρέας Μέλτσα για 1,5 λεπτό. Εν Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όλοι γνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι ε, θεωρούν την Ευρώπη ε, σαν ένα γραφειοκρατικό τέρας ε, το οποίο λαμβάνει αποφάσεις πάνω από τα κεφάλια του λαού. Η διοίκηση της, των Βρυξελών θα έπρεπε να έχει μειώσει το έργο της και να έχει αυξήσει τη διοίκηση διαφάνεια και αντί να μιλάμε για μία επανεθνικοποίηση ε, και να υπερβάλλουμε ε, πρέπει να αντιληφθούμε ότι ε, οι αρμοδιότητες των κρατών είναι να είναι και υπόλογοι προς τους πολίτες. Καλό λοιπόν θα ήταν να έχουμε μειώσει όλη αυτή τη συγκέντρωση και να κοιτάξουμε να προωθήσουμε την συνεργασία για την μείωση της παράνομης μετανάστευσης. Ε, βλέπουμε ότι στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως υπήρχε ξεμία μεταβολή προς μία Ευρώπη χρεών και ε, ε, πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ διότι βλέπουμε ότι η Δανία έχει μεταφέρει χρονικά το δημοψήφισμα για μια μεγαλύτερη εμπλοκή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τελικά όλες οι προσπάθειες αποδειχθούν χωρίς αποτέλεσμα εφόσον υπάρχει μια Ευρώπη των χρεών. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να εκφράσω ειλικρινή συγχαρητήρια στην Δανέζικη Προεδρία για την εξαιρετική της εργασία και για τα σημαντικά αποτελέσματα που επέτυχε στη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Εξαμένου. Θα ιδιαίτερα να σας συγχαρώ για τις διαπραγματευτικές σα ικανότητε, τι εξαιρετικέ που συνέβαλαν στην ολοκλήρωση ε, μάλλον στην αποφυγή της ολοκλήρωσης αυτής της ε, παράλογης συμφωνίας ε, για τα, τις ευρεσιτεχνίες. Επίσης, αναβολή της μονομερούς πρότασης του Συμβουλίου για την πρόταση κανονισμού. Ε, δεν μπορώ ωστόσο να μην τονίσω ότι σοβαρά επηρεάζεται η ισορροπία η θεσμική της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυρίως για ένα θέμα το οποίο είναι τόσο σημαντικό για την πρόθεση της ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης της δομής κλειδιά όπως η καινοτομία. Υπάρχουν διατάξεις όπου το Κοινοβούλιο είχε την προγραμματική και επικοδομητική θέση. Γι' αυτό και εκφράζω την πικρία μου για τα όσα συνέβησαν και καλό το Συμβούλιο των Υπουργών που εκπροσωπείται από την ε, Κυριακή Προεδρία να βρει θέσεις ε, διαφορετικές για τη δημοσία και για την διαδικασία. Το Κοινοβούλιο ε, δεν θέλει να προκαλέσει την αποτυχία ενός προγράμματος ε, που έχει διαρκέσει εδώ και 30 χρόνια, ούτε το Κοινοβούλιο θα επιτρέψει η πειθαρχία και οι θεσμικές σχέσεις να αντιστρέφονται κατά βούληση. Φερνάντο Λόπεθ, Ακιάρ, για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρωθυπουργέ. Η Προεδρία της Δανίας ήταν φορτωμένη με πάρα πολύ υψηλές προσδοκίες, ε, με μια κυβέρνηση η οποία έπρεπε να μπει μέσα σε αυτό το αγώνα για την κρίση. Όμως δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι όταν κάνουμε την αξιολόγηση και έχουμε επίσης και την ε, ε, απόφαση του να ε, ξαναγυρίσει το Σέγγεν στα χέρια της, των κρατών μελών. Επομένως, έτσι αγνοούμε αυτό τον κοινό χώρο δικαιοσύνης και ασφάλειας εμείς εκεί είμαστε συνομοθέτες ξέρετε ως κοινοβούλιο γιατί έχουμε τώρα το Σέγγεν το οποίο αφορούσε μισό 500 εκατομμύρια Ευρωπαίους και οπότε στην Κοπενχάγη αυτό το οποίο καταφέρατε είναι να αγνοήσετε το άρθρο 80 για την αλληλεγγύη γιατί έτσι ε, τώρα τι θέλουμε να βάλουμε ξανά ε, να, κάνουμε, να, βάλουμε, να βάλουμε ξανά εσωτερικά σύνορα ενώ, ενώ αυτό το οποίο θέλουμε σε αρχή να έχουμε κοινή διαχείριση των κοινών σύνορων οπότε επ' αυτού έχω να σας πω ότι αυτό αφορά όλο το Σέγγεν και όλο το, το, τις ρυθμίσεις για το Άσυλο και για το Σέγγεν όμως τι λέτε, τι λέτε εσείς για τις εγγύησεις των, των καταθέσεων, τι λέτε για το πακέτο για τις τράπεζες, εκεί θα πρέπει να επιδειχθεί αλληλεγγύη. Γεράρ, ε, δέχεστε μπλε κάρτα από τον κύριο Λόκεγκάρτ. Κύριε Λόκεγκάρτ. Κύριε Λόκεγκάρτ. Ε, Λόκεγκάρτ. Ευχαριστώ. Και εγώ με την ευκαιρία να σας αναφέρω κάτι. Θεωρώ ότι πέτυχε η Προεδρία της Δανίας. Ευχαριστούμε για την τόσο θετική συνεργασία, αλλά αυτό το οποίο με πείραξε είναι ότι η Προεδρία δεν εστίασε την προσοχή της περισσότερο στο τι θα γίνει μετά την κρίση. Πώς θα ανακτήσουμε την δημοκρατική νομιμότητα ε, στα μάτια των πολιτών. Okay. Μπλε κάρτα σημαίνει ότι απευθύνεται ερώτηση στον προλαλήσαντα συνάδελφο. Δεν είναι διαδικασία catch the eye, εκτός και αν σηκώσατε λάθος ε, κάρτα. Έχετε κάποια ερώτηση προς τον κύριο συνάδελφο, τον προλαλήσαντα, τον κύριο Λόπεθ Αϊλάρ. Όχι, αυτό ήταν ε, παρατήρηση για την Προεδρία. Αν δεν γίνεται τώρα, το πω Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Επόμενος ε, ομιλητής είναι ο κύριος ε, Κάλφιν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρωθυπουργέ, θα ήθελα να σε χαρώ και να ευχαριστήσω τη Δανέζικη Προεδρία και ιδιαίτερα στον Υπουργό Βάμεν γιατί αντιμετώπισαν ένα από τα πιο δύσκολα και ευαίσθητα ντοσιέ. Δηλαδή το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Ξέρω ότι υπάρχουν πολλέ αντιφάσει, αλλά τόσο συνέβησαν κατά τη διάρκεια της Δανικής Προεδρίας ε, οδήγησαν σε ευθυγράμμιση τη συζήτηση για, ε, δημιούργησε τις προϋποθέσεις για μια ε, πιο εύκολη συμφωνία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητήθηκε, ε, συζήτησε περισσότερο το θέμα. Θα ήθελα περισσότερα αποτελέσματα ωστόσο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την πολύ καλή διαθεσμική συνεργασία. Δόθηκε πρώτη φορά, στην πρώτη φορά στην ευκαιρία να μιλήσει το Κοινοβούλιο με το Συμβούλιο και να δώσει ε, τις απόψεις του για το πολιετές πλαίσιο και επίσης ε, να συγχαρώ την Προεδρία για τα συμπεράσματα. Πιστεύω τα όσα πετύχατε ήταν πολύ καλή βάση για συμφωνία για το ΠΔΠ. Ευχαριστώ. Διαδικασία Catch the Δίνω το λόγο στη συνάδελφο κυρία Γκρέσλε.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 Κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε του Συμβουλίου, σαν μέλος της Επιτροπής Υπολογισμού, θα ήθελα να σας πω ότι αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μία διαδικασία για τη δημοσιονομική περίοδο. Η διαδικασία της Όλαφ είναι στο Συμβούλιο πολύ καιρό και μπορέσατε να την ολοκληρώσετε γι' αυτό θέλω να σας ευχαριστήσω όπως να ευχαριστήσω και τους υπαλλήλους οι οποίοι επεξεργάστηκαν τον τομέα αυτό και το φάκελο αυτό διότι εξυπηρέτησαν τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και σας ευχαριστώ. Λόγω έχει τώρα η συνάδελφος κυρία Γκουρμάη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε ε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, πριν έξι μηνών είχα πει ότι έχουμε μεγάλες προσδοκίες από τη Δανική Προεδρία, όχι μόνο διότι ηγείται γυναίκα, αλλά διότι υπάρχουν πολλές προκλήσεις για την Ευρώπη. Έξι μήνες είναι λίγος χρόνος για να ανταποκριθεί κανείς σε αυτές τις προσδοκίες. Πιστεύουμε όμως κατόπιν του τελευταίου Συμβουλίου ότι αν υπάρχει ε, ομόνια πολλά μπορούν να επιληθούν, να επιληθούν. και αναφέρομαι εδώ εις ε, τη ε, φόρο δημοσιονομικών συναλλαγών και θέλω να ευχαριστήσω την Προεδρία και ιδιαίτερο τον κύριο Μπάμεν για την εργασία τους ιδίως στο θέμα της ισότητας των φύλων σε πολλά θέματα προχώρησαν πολύ αλλά ακόμη δεν υπάρχει συμφωνία σχετικά με την οδηγία για την άδεια μητρότητος. Πρέπει λοιπόν να αναλάβουμε τις ευθύνες μας, να μην εγκαταλείψουμε το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο και σας ευχαριστώ. ο Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό για την Πρωθυπουργό για την εξαιρετική εργασία κατά τη Δανική Προεδρία. Ελπίζω ότι αυτό θα συνεχιστεί και βεβαίως ότι θα υπάρχει πρόοδος και στο μέλλον. Με τα χαράς διαπίστωσα ότι μπορέσαμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία σχετικά με το κόστος για τη χρέωση της περιαγωγής και στη, σχετικά με την οδηγία για την εξοικονόμηση ενεργείας. Βεβαίως ε, ε, ε, η Ιρλανδία θα αναλάβει την Προεδρία στην αρχή του 2013 και ελπίζουμε ότι κατά την δικιά μας Προεδρία θα επιτύχουμε όσα επέτυχε και η Δανία. Και πάλι ευχαριστώ τη Δανία. σε ευχαριστώ. Θα ξαναπροσπαθήσω. Όπως έλεγα πριν από λίγο, θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, Δανέζικη Προεδρία την οποία εκτιμάμε ιδιαίτερα καθώς και σε τον ε, Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ε, κύριο Βάμεν. Το τελευταίο εξάμενο έγινε μια συζήτηση στην Ευρώπη που στηρίχθηκε κυρίως από τη Γερμανία για το πώς θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε πώς θα μπορέσουμε να έρθουμε πιο κοντά στους ε, λαούς μας. Ίσως η Δανέζικη Προεδρία να μην συμμετείχε πολύ ενεργά. Θα μπορούσε να έχει εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία ευκαιρία και να συνεργαστεί πιο συγκεκριμένα με το Ευρωκοινοβούλιο για να προωθήσει τη συζήτηση. Andrew Bronz. Those who advance the European project see themselves as Όσοι ε, θεωρούν ότι προχωρεί το ευρωπαϊκό πρόγραμμα θεωρούν τους εαυτούς τους ως ευρωπαϊστές. Ωστόσο αυτό οδεύει προς καταστροφή και αυτό μπορεί κανείς να το δει σαφώ στο πρόγραμμα της Δανέζικης Προεδρίας. Η Δανία προσπάθησε να προχωρήσει και να προωθήσει την υποψηφιότητα της Τουρκίας που, μιας χώρας που πατροπαράδατα και πολιτιστικά δεν είναι ευρωπαϊκή. Προσπάθησε να σταματήσει την παράνομη μετανάστευση, ε, μάλλον να ε, διευκολύνει την μετανάστευση, την, παρά, την νόμιμη ε, ισχυριζόμενοι πως χρειαζόμαστε περισσότερους μετανάστες εδώ, με γραφειοκρατική πρόσβαση λέει. Ε, επίσης είπε πολλά λόγια για την επιστροφή των παράνομων ε, μεταναστών. Ξέρουμε από τη Frontex ότι δεν κρατούνται επί μακρόν, αλλά τους δίνεται δίθεν η εντολή να φύγουν, αλλά κανένας δεν ελέγχει αν εφαρμόζεται η εντολή. Οι λαοί της Ευρώπης δεν, μπο μπορεί εύκολα να αντικατασταθούν από ανθρώπους από τον τρίτο κόσμο. Ευχαριστώ η κυρία Γιακοψάρη. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θεωρώ ότι ίσως ο κόσμος αναρωτιέται Πώς είναι τον εδώ να αλληλοσύγχερόμεθα ενώ η αγορά είναι έξαλλη για τα χτυπήματα που δέχεται από την κρίση. Εγώ νομίζω ότι η συνάντηση κορυφής ήταν ένα ναυάγιο. Ήταν τρομερό το να ακούει κανείς τους ε, ε τα μέλη τους εκπρόσωπων των μελών τέλος πάντων να τα λένε μεταξύ τους ε, ήταν, ήταν αποτρόπη η κατάσταση. Είδαμε τι έγινε και με το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. τόσο τόσε, τόσε σημαντικές αποφάσεις ελήφθησαν ε, διανυκτός τότε, στην και το θέμα είναι ότι κανένας έχοντας ξενυχτήσει τόσο πολύ ε, είναι σαν ένας μεθυσμένος να προσπαθεί να οδηγήσει. Δεν θα πρέπει να λαμβάνονται αποφάσεις υπό τέτοιε συνθήκες ξενυχτιού, διανυκτός. Τι λέτε κυρία Πρωθυπουργέ, πώς είναι δυνατόν να έχουμε τέτοια πράγματα, πώς θα το αποφύγουμε στο μέλλον. Ε, din păcate, președinția daneză a fost ε, umbrită de criza instituțională fără Ε, περάσαμε μια θεσμική κρίση άνευ προηγουμένου μέσω της, απο, του, αποκλεισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από την συστήμα αξιολόγησης του Σέγγεν. Άμεση απίπτωση δε του συστήματος αυτού στους Ευρωπαίους πολίτες και μάλιστα σε μια εποχή μετά τη Λισαβόνα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έπρεπε να, μείνει σε, να, να, να κρατηθεί σε απόσταση όταν λαμβάνονται τόσο σημαντικές αποφάσεις. Η Δανία παραδοσιακά ψήφισε υπέρ διαφάνειας ε, των αποφάσεων. Όμως με αυτή την απόφαση ο υπολογισμό μας για την Προεδρία σα δεν μπορεί να είναι μόνο θετική. Εκφράζω την ευχή η Κυπριακή Προεδρία να μπορέσει να φέρει σε αίσιο πέρα σε αυτή τη διαδικασία με πολλά περισσότερα θετικά στοιχεία για το Κοινοβούλιο και εμπλέκοντάς το στη ε, διαδικασία λήψη αποφάσεων ολοκληρώθηκε η διαδικασία κάτω τώρα και το λόγο έχει ο κύριος Ζεφ Ζεφκοβιτς εν ονόματι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αγαπητέ, αγαπητή κυρία Πρωθυπουργέ, αγαπη, ε, Πρόεδρε, ε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτέ, αυτή η πλούσια συζήτηση έδειξε αυτό που αναφέρθηκαν από διάφορου ομιλητέ, ότι η Δανέζικη Προεδρία δούλεψε σκληρά δυναμικά, πρακτικά και επέτυχε πολλά και σε πολλά μέτωπα η πρόοδος ήταν ε, σαφής και εμείς το εκτιμήσαμε ιδιαίτερα. Παρά τις προσπάθειες είναι σαφές ότι για την ενέργεια και την ότι την ενεργειακή απόδοση ε, το Σέγγεν ε, θα έχουμε περισσότερες προσπάθειες να κάνουμε. Χρειάζεται περισσότερη φιλοδοξία και σεβασμό στην κοινωτική μέθοδο. Ιδιαίτερα εκτιμώ τις προσπάθειες της Δανικής Προεδρίας και τα αποτελέσματά της καθώς και τον τρόπο με τον οποίο έγιναν οι συζητήσεις και οι διαπραγματεύσεις για το πολυμερές δημοσιονομικό πλαίσιο. Η Προεδρία σας ε, οδήγησε στο διαπραγματευτικό ε, κούτι μια καλή βάση επί της οποίας μπορούμε όλοι να δουλέψουμε ώστε να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις μέχρι το τέλος του έτους. Ήσασταν σαφείς όσον αφορά τη σημασία της στενής συνεργασίας με την αντιπροσωπεία ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιου. Συνεχίσατε τακτικές συνεντήσεις που σίγουρα θα στρώσουν το δρόμο για αυξημένη συνεργασία ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε με αυτές τις σημαντικές ε, συνομιλίες μέχρι το τέλο του χρόνου. Επίση να τονίσω ότι ε, άνοιξε και το διαπραγματευτικό κουτί με το Μαυροβούνιο ε, για την ένταξη ανοίγοντας, δίνοντας μάλλον το καθεστώς υποψήφιου κράτους στην Σερβία και ανοίγοντας έτσι το δρόμο για διαπραγματεύσεις και με τα άλλα βαλκανικά κράτη. Τέλος να ευχαριστήσω ε, για την προσωπική του προσήλωση τον Υπουργό Βάμεν που με βοήθησε να επιτύχω πρόοδο στο εφάκελο που ήταν στο πιτάπιτος εδώ και τρία χρόνια δηλαδή πώς θα διαχειριστούμε καλύτερα ε, τους οργανισμούς στο μέλλον. Έχουμε δουλέψει πολύ σκληρά υπό την με την αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από την προεδρία τη κυρία Γιούτα Χάουγκ και είμαι πεπισμένο απόλυτα ότι η κοινή μα προσέγγιση επί των αρχών θα μα βοηθήσει να αποφύγουμε καταστάσει όπω αυτέ που αντιμετωπίζουμε με το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρυστεχνία και θα μπορέσουμε να χειριστούμε και τη συζήτηση για τα όσα θα χρειαστεί να φτιάξουμε στο μέλλον οργανισμούς δηλαδή με πολύ πιο αποτελεσματικό και οργανωμένο τρόπο. Σας ευχαριστούμε πολύ Πρόεδρε που μας δώσατε το λόγο και ευχαριστούμε τη Δανέζικη Προεδρία για τη μεγάλη της προσπάθεια και τα σπουδαία αποτελέσματά της. Ευχαριστώ κύριε Ζεύκοβιτς. Δεν ξέρω τι ήταν ο θόρυβος ο οποίος ε, έγινε. Ελπίζω ότι δεν συνέβη κάτι δυσάρεστο. Ευχαριστώ λοιπόν κύριε Ζεύκοβιτ. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Τόνι Σμιτ. Και πάλι κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων και αξιότιμοι κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές. Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω για τα καλά σας λόγια και δύο προς τον Νίκολα Μπάμεν, τον ε, Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, διότι είναι πολύ ε, μεγάλη χαρά που εκτιμήσατε την ε, σκληρή δουλειά την οποία οποία έκανε. Σημείωσα τις παρατηρήσεις σας και είδα ότι έχουμε την κοινή προσήλυση να φέρουμε την Ευρώπη στο σωστό δρόμο και να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίες για του τόσους πολλούς ανέργους. Ε, αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε σε μία δύσκολη περίοδο στην Ευρώπη και χάρη στην εργασία αυτού του Κοινοβουλίου καταφέραμε να κάνουμε μεγάλες προόδους προς αυτή την κατεύθυνση Τώρα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα συνεχίσουμε από κοινού να δημιουργούμε και να υλοποιούμε τους στόχους μας και μέσω του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου διότι οι πολιτικοί μας και οι πολίτες μας βλέπουν και περιμένουν από μας νέες θέσεις εργασίας και νέα πρόοδο και ανάπτυξη. Πρέπει δε αυτό να γίνει με εφαρμογή της κοινοτική μεθόδου. Τι σημαίνει αυτό, ότι πολλές φορές συζητάμε και τσακωνόμαστε σχετικά με τα οράματα του καθενός και έτσι έχει γίνει στο παρελθόν έτσι έγινε και στη δανική περίοδο της Προεδρίας αλλά δεν πρέπει να ανησυχούμε πολλές φορές πρέπει να φτάσουμε σε συμβιβασμούς άλλοτε συμφωνούμε άλλοτε όχι αλλά όλον ο κοινό στόχος είναι να εξυπηρετούμε τους πολίτες θέλω τώρα να αναφερθώ σε ορισμένα θέματα τα οποία συζητήσατε σήμερα πολύ σωστά είπατε ότι ακόμη είμαστε σε πολύ κακή οικονομική κατάσταση και σε μεγάλη κρίση και έτσι είναι και αυτό θα συνεχιστεί για κάποιο χρονικό διάστημα. Κάθε μέρα έχουμε ε, μία νέα επίπτωση της οικονομικής ε, κρίσεως και χιλιάδες ανέργους στην Ευρώπη. Γι' αυτό και χαίρομαι τόσο πολύ ότι πολλοί από εσά συμμερίστηκαν την ανησυχία μου να προωθήσουμε το Σύμφωνο Ανάπτυξης και Απασχόλησης διότι για δεν αρκούσε αυτό το σύμφωνο αλλά θα συμφωνήσετε ότι τουλάχιστον είναι ένα φως στο σκοτάδι που θα δημιουργήσει κάποια ελπίδα ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε και πάλι θέσεις εργασίας στην Ευρώπη. Το συζητήσαμε και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την Πέμπτη και την Παρασκευή και όπως σας είπα δεν ε, είχα κανένα δισταγμό να συστήσω στο Συμβούλιο να ενισχύσουμε τη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα πλαίσια αυτά για να δημιουργήσουμε δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας και να μπορέσουμε ενδεχομένως να προωθήσουμε ορισμένες από τις αποφάσεις που έπρεπε να ληφθούν. Σε κάθε βήμα πρέπει ε, να σεβόμαστε τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ε, αυτό είναι πλήρη συνείδηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και όλοι θέλουμε να μπορέσουμε να αποδώσουμε ε, το σύμφωνο αυτό γιατί αυτό περιμένουν και οι πολίτες της Ευρώπης από μας. Θέλω να ευχαριστήσω αυτούς που αναφέρθηκαν στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και να ευχαριστήσω και όσους από εσάς συμμετείχατε στο Κοινοβούλιο στη συζήτηση αυτή. Ο διάλογος ήταν επικοδομητικός όπως και οι απραγματεύσεις που είχαμε στη, κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σε όλα τα επίπεδα. Προσπαθήσαμε να σεβαστούμε το παρελθόν του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να τονίσουμε από την πρώτη μέρα τις απόψεις και να τις προβάλλουμε στις συζητήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Νομίζω ότι ήταν η πιο στενή συνεργασία επί του θέματος αυτού μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Ελπίζω δε ότι η εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα μπορέσει να συνεχιστεί εξίσου επικοδομητικά όπως ξεκίνησε από εσά αναφέρθηκαν στα διπλώματα ευρεσιτεχνία και στο σχετικό κανονισμό και σημείωσα τι παρατηρήσει σα σχετικά με, τις, ε, ε, με τα διπλώματα ευρεσιτεχνία. Μην ξεχνάτε ότι η Ευρώπη περιμένει 30 χρόνια τη λύση και όταν περιμένετε 30 χρόνια ξέρετε ότι η λύση θα ε, χρειαστεί κάποιο συμβιβασμό. Αντιλαμβάνομαι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεχίσει τη συζήτηση αυτή το Σεπτέμβριο και ελπίζω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορέσει να αναλάβει τις ευθύνες του και να καταλήξουμε σε μια τελική συμφωνία για τη διατήρηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης στην Ευρώπη. Ξέρουμε ότι ορισμένοι έχουν διαφορετικούς στόχους, ξέρω τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά σας απευθύνω μία έκκληση να μην καταλήξουμε σε μία κατάσταση και να μην γίνει το βέλτιστο εχθρός του καλού. Ένα άλλο θέμα το οποίο χάρηκα πολύ κατά τη συζήτησή μας σήμερα ήταν οι πολλές παρεμβάσεις σχετικά με ε, το πράσινο πρόγραμμα διότι ξέρετε ότι δεν ήταν εύκολο να προωθήσουμε το πράσινο πρόγραμμα σε ε, ε, μία περίοδο κρίσεως αλλά είμαι πολύ ε, ικανοποιημένοι με την ε, επιτυχία μας ιδίως όσον αφορά την πράσινη αποτελεσματικότητα και χάρη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον πρόεδρό της κύριο Μπαρόζο μπορέσαμε να προωθήσουμε την πράσινη οικονομία έγινε αυτό κατά τη διάρκεια των έξι μηνών ο κύριος Μπαρόζο το προώθησε και ξέρω ότι θα συνεχίσει να το προωθεί η προσήλωση του κυρίου Μπαρόζο είναι σημαντική και ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτό και ε, προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του σήμερα και του αύριο. Η κρίση που υπάρχει αυτή τη στιγμή και οι λύσεις που βρίσκουμε δείχνουν ότι ακόμη και αν δεν συμφωνούμε πάντοτε δεν πρέπει να απελπιζόμαστε. Πρέπει να είμαστε αλληλέγγυοι και να συνεχίσουμε να την επιδεικνύουμε να επιδεικνύουμε την αλληλεγγύη αυτή ε, διότι όλοι αντιμετωπίζουμε σοβαρή κρίση αλλά οι αποφάσεις οι οποίες παίρνουμε από κοινού θα μας οδηγήσουν σε μία διέξοδο από την κρίση και σε ένα καλύτερο μέλλον. Ελπίζω ότι θα κριθούμε βάσει τις δυνατότητές μας να συνεργαστούμε, να βρούμε συμβιβαστικές λύσεις και οι ηγέτες σήμερα αποφασίζονται από τα αποτελέσματα και όχι από τις προθέσεις. Αυτό το οποίο περιμένουμε περιμένουν οι Ευρωπαίοι από εμά είναι αποτελέσματα, λύσεις και προσπαθήσαμε να ανταποκριθούμε σε αυτή την υποχρέωση κατά το τελευταίο εξάμεινο και θα συνεχίσουμε το πράττουμε και στο μέλλον κατά τρόπον ώστε η Ευρώπη να ξεφύγει από την απεσιοδοξία και να προσβλέπει προς ανάπτυξη και αισιοδοξία και αυτό είναι δυνατόν μόνο εάν δεσμευτούμε ότι θα το πράξουμε από κοινού και σας ευχαριστώ για τις συνεργασία σας. Ευχαριστώ κυρία Πρωθυπουργέ για τα λόγια σας. Κυρίες και κύριοι, η συζήτηση του απολογισμού της Δανεικής Προεδρίας τελείωσε. Θα έχουμε ένα μια σύντομη διακοπή. So. Herr Minister Wammen, ich Wammen, Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ. Ε, ε, ε, άντε, γεια σου, γεια σου, Νικολάη. Κυρίες και κύριοι, σας παρακαλώ να πάρετε πάλι τις θέσεις σας και θα συνεχίσουμε τη συζήτηση.